συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση. Έχετε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνονται τα πρακτικά. Το επόμενο σημείο